αυτή την ημέρα της, που είναι η διεθνή ημέρα κατά τη μορφή αυτής βίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ο λόγος στην κυρία Κοράτσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επιτροπέ, φίλε. Είναι καλό που σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας ασχέτως ε, πολιτικής ε, προέλευσης με μεγάλη συνένεση, με μια ισχυρή έκκληση για να σταματήσει αυτή η βάρβαρη πρακτική του εκοτηρισμού των γυναικείων γενετικών οργάνων. Καλωσορίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναλαμβάνει δέσμευση με την ανακοίνωσή τη να προσθέσει δράσει και χρηματοδότηση στον εντοπίση του φαινομένου αυτού. Ήδη αναφέρθηκαν οι αριθμοί που πραγματικά ε, μα ε, δημιουργούν, ε, μα προκαλούν πόνο. Μιλάμε για εκατομμύρια γυναίκε, παιδιά, κοριτσάκια. Ακόμα και μέσα στην ίδια την Ευρώπη έχουμε μισό εκατομμύριο γυναίκε που κινδυνεύουν. Ε, μπροστά μας. Οπότε το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε ως μια μορφή βίας κατά των γυναικών, ως μια μορφή βίας κατά των παιδιών. Θα πρέπει να υπάρξουν ποινικέ συνέπειες, καλό τα κάτι μέλη, να αντιμετωπίσουν τον εκατηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως έγκλημα και να αυξήσουν τα μέτρα πρόληψης αλλά και την δίωξη την, ε, του φαινομένου αυτού λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις και τις αξίες της σε άλλου άλλους πολιτισμούς με διαφορετικές παραδόσεις. Αυτό το θεωρώ απαράδεικτο, διότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Αθηνών Μπανκιμούν είπε ο ίδιος ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα, τις μεγαλύτερες ε, πολιτιστικές αξίες που έχει ο κάθε πολιτισμός και να αφήσουμε τα αρνητικά πίσω μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την ε, ε τόλμη να πούμε ότι δεν μπορεί η βία να δικαιολογείται από την παράδοση, την ιστορία, τη θρησκεία. Ε, όχι, ψάχνουμε οικουμενικές αξίες που έχουν ε, ήδη καταγραφεί ούτως ή άλλως στην ε, Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς προς αυτό. Επίσης, θα πρέπει η πολιτιστική, μάλλον η κουλτούρα ως προς τα θέματα αυτά, η νοοτροπία να αλλάξει και να υπάρξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, για τα δικαιώματα των γυναικών. Όπως προσπαθεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και πολλές ενώσεις των γυναικών στα κράτη-μέλη μας. Πρέπει να συνεργαστούμε με επαγγελματίες σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η πρόληψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να εντοπίσουμε καλύτερα τις ομάδες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και να μπορέσουμε να προσφέρουμε πρόληψη, μέτρα πρόληψης Πρόεδρε, εγώ συμμετείχα στην εκστρατεία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μηδενική ανοχή κατά του ακροτηριασμού των γυναικείων γενετικών οργάνων και ελπίζω ότι όλοι θα δεσμευτούμε στον αγώνα αυτό και θα ε, επιδιώξουμε μαζί έντονη δράση. Ε, πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Παρόλο το, παρά το γεγονό ότι το φαινόμενο αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο από τη Διεθνή Κοινότητα Υγεία και του ε, εντυπωσιακού αριθμού, το φαινόμενο παραμένει ενισχυτικό εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για σοβαρή παραβίαση των, κατάφορη παραβίαση των ε, βασικών δικαιωμάτων ε, γυναικών και κοριτσιών, αλλά πραγματικά θέτει σε κίνδυνο